ευχαριστώ και τον Επίτροπο Έτσιγκερ καλώς καθώς και τους εισηγητές που έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή, που ολοκληρώνεται εδώ. Και τώρα περνώ στο δεύτερο θέμα της ε, απογευματινής μας συνεδρίασης. Έκθεση της κυρίας Βαλέρο, έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων, εφαρμογή της κοινή θέση 2008. 944 και θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαλέρο για 4 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ τους και ηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο θέμα αυτό, στην έκθεση αυτή. Μπορεί να μην συμφωνήσαμε σε όλα, αλλά είμαι βεβαία ότι συμφωνούμε ως προς το τι εννοούμε ε, και ως προς τον στόχο του ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Όταν δηλαδή ε, λέμε ότι δεν πρέπει τα όπλα να καταλήγουν σε λάθος χέρια, ακόμα και να έχουμε διαφορετική αντίληψη σχετικά με άλλα πράγματα, συμφωνούμε όλοι. Είναι ένα θέμα λοιπόν και εσωτερικό αλλά και εξωτερικό, εξωτερικού εμπορίου, εξωτερικής πολιτικής στο θέμα των εξάγων όπλων. Εσωτερική πολιτική καθίσταται όταν βλέπουμε τρομοκράτες να διαπράττουν τις ε, φωνικές τους επιθέσεις με όπλα προερχόμενα από ευρωπαϊκές εξαγωγές. Είδαμε ότι αυτό συνέβη στη Βαρκελόνη. Μάλιστα μάθαμε ότι ο Ισπανός ε, ε, βασιλέα σκοπεύει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία για να συζητήσει ακριβώς το θέμα των εξαγωγών των όπλων. Ζητούμε ε, να συζητηθεί ανοιχτά το θέμα της ειρήνης, ε, τα όπλα που πηγαίνουν Σαουδική Αραβία η οποία και χρηματοδοτεί τεμένη αλλά και βοηθεί με τον τρόπο της την ρουσπαστικοποίηση ορισμένων που επισκευούνται αυτά τα τεμένη στην Ευρώπη έχει ευθύνη ως προς την ε, τρομοκρατία. Προσφέρει επίσης όπλα στην ε, Αλνούστρα, την Αλκάιντα, την Ίσης η Σαουδική Αραβία και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ευρωπαϊκά όπλα να καταλήγουν στα χέρια αυτών των τρομοκρατών. Έχουμε λοιπόν μια κοινή θέση με 8 σημεία κανονισμό ε, ο οποίος είναι σαφέστατος και ε, ξεκάθαρος ως προς το που μπορούν να εξάγονται τα όπλα, γιατί δεν επιτρέπεται να εξάγονται σε ε, χώρε που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, τα κριτήρια δεν εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη. Εάν συνέβαινε αυτό, εάν τα κράτη-μέλη εφάρμοζαν σωστά τα ε, κριτήρια, τα κράτη-μέλη, δεν θα έπρεπε κανένα όπλο ευρωπαϊκό να φτάνει στη Σαουδική Αραβία. Επειδή όμω ερμηνεύουν διαφορετικά τον κανονισμό από ό,τι θα όφυλαν τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ε, αυτά τα προβλήματα. Έχουμε επίση κράτη τα οποία ενδεχομένω έχουν αγοράσει όπλα ή λοιπόν στρατιωτικό εξοπλισμό σε περίοδου ειρήνη που όμως έχουν εντωμεταξύ εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις σε άλλες χώρες ή υποστηρίζουν ε, με, τον, με την παροχή αυτών των όπλων και εξοπλισμών ε, ένοπλες ε, ομάδες σε άλλες χώρες. Πώς μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε, αυτή τη ροή δηλαδή των όπλων και την μεταπόλησή τους είναι κάτι το οποίο δεν, μπορεί, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όπως έχει τώρα η κατάσταση αλλά έχουμε καλέσει ως Κοινοβούλιο στην επιβολή ενός εμπάργου ε, απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και άλλα μέσα έχουμε ζητήσει να αναπτυχθούν αλλά πάντως ε, το εμπάργο είναι ένας απαραίτητος ε, όρος για χώρα η οποία παραβιάζει τους κανονισμούς μας και επίσης πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο πιθανή χρήση του εξοπλισμού που εξάγεται αλλά και ποια είναι η κατάσταση στη χώρα στην οποία εξάγονται τα προϊόντα, πώς διατίθενται οι άδειες και ποια είναι η κατάσταση στην εποχή που έχουν από την εποχή που έχουν διατεθεί μέχρι την εποχή που ε, υλοποιούνται οι εξαγωγές. Επίσης είναι δυνατόν να έχουμε ένα τόσο μεγάλο δυναμικό παραγωγής όπλων στη χώρα μας, στις χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τόσο μεγάλο ποσοστό των όπλων μας να φτάνει μέσω των εξαγωγών στη Μέση Ανατολή και μόνο 15% των, οπλικών μας, ε, ε, των όπλων και των οπλικών συστημάτων να ε, εξάγεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτά τα επίπεδα παραγωγής όπλων, δεν μπορούμε να, να επικαλούμε θα καν ε, την έννοια της διαφύλαξης θέσεων εργασίας στην παραγωγή και εξαγωγή όπλων. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε την εξαγωγή όπλων προς χώρες οι οποίες παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε πιο αυστηρούς ελέγχους λοιπόν, θέλουμε κυρώσεις προς τις χώρες οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες και θέλουμε κυρία Μογκερίνη το, ε, το φύλλο της, ε, του εμπάργου, το επιχείρημα και το μέσον πιέση που είναι το εμπάργο, να το χρησιμοποιεί κάθε φορά και εδώ μιλούμε όχι μόνο για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά και για τη ζωή και την ασφάλεια των δικών μας πολιτών. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο, ο Υπουργός κ. Μαζίκας είναι εδώ και τον καλωσορίζουμε. Εξ ονόματος ε, δε της ε, Ευρωπαϊκής... Ε, και θα μιλήσει εκ μέρους κυρίας κυρία Μογκερίνα, την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη, στο όνομα της ε, εκπροσώπου μιλάω, της κυρίας Μογκερίνη ε, και καλωσορίζω αυτή την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση αλλά και την προπαρασκευή και την συζήτηση της έκθεσης που προετοίμασε η κυρία Βαλέρο είναι ένα ζήτημα που αφορά κοινοβουλευτικό έλεγχο σε ό,τι αφορά την ε, πώληση όπλων και σχετίζεται με το θέμα της διαφάνειας γενικότερα. Τα ζητήματα αυτά της εξαγωγής όπλων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον ακαδημαϊκό κόσμο, με την κοινή γνώμη, έχουν ε, αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Δείχνει ότι η διαφάνεια και ο διάλογος μπορεί να, γίνει χώρα, να λάβει χώρα χωρίς να ε, θίγονται οι ευθύνε και αρμοδιότητε των εμπλεκόμενων φορέων. Ε, ζητούμε μεγαλύτερη διαφάνεια παγκοσμίω μέσω της ε, συμφωνίας για την εμπορία όπλων. Η διαφάνεια όμως δεν πρέπει να αντιβαίνει την, εθνική, την εθνική και την περιφερειακή ασφάλεια. Υπάρχει μια κοινή θέση της Ένωσης που έχει πάρθει το 2008 υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή το οποίο ενιαίο βασίζεται στην εθνική ευθύνη για την πώληση όπλων ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Η ευρωπαϊκή κοινή θέση σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ό,τι αφορά το, το, το ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι σαφής και βεβαίω υπάρχει το θέμα της επίπτωσης στην εσωτερική και τη διεθνή σταθερότητα. Η αδειοδότηση ό,τι αφορά την ε, πώληση όπλων διέπεται από έναν οδηγό ο οποίος ε, έχει μεταρρυθμιστεί το 2015. Υπάρχει λοιπόν μια εθνική ευθύνη η οποία ασκείται με κοινά κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου. Ο συνολικό στόχο τη κοινή θέση τη Ένωση είναι να προωθήσουμε υπεύθυνε πολιτικέ πώληση όπλων και σύγκληση. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το Συμβούλιο και η Υπηρεσία εξωτερική δράση ε, έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχει και ομάδα εργασία του Συμβουλίου για την εξαγωγή όπλων καθώ και μια πλατφόρμα IT που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση κινδύνου με λεπτομέρειε ό,τι φορά τι αρνήσει αδειοδότηση Όπω και δύο γραμμέ, αυτή Αυτές ε, οι δυνατότητες αλλαγής πληροφοριών έχουν επικαιροποιηθεί πρόσφατα μετά την αναθεώρηση της κοινή θέση της Ένωσης που επετεύθη το 2015. Αυτό εξακολουθεί να συνεισφέρει στην σύγκληση των πολιτικών πώλησης όπλων καθώς αυτές ε, εφαρμόζονται. Τώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γειτονιά μας, μια σειρά από τρίτες χώρες έχουν ευθυγραμμιστεί με τα κριτήρια της κοινή θέση της Ένωσης. Για να τους βοηθήσουμε στην καθημερινή επιχειρησιακή εφαρμογή, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα προ... πρόγραμμα ε, συνεργασίας και προσέγγισης. Το τελευταίο πρόγραμμα για την περίοδο 2016-2017 θα λήξει το Δεκέμβριο. Όμως ήδη έχουμε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί το πρόγραμμα και για τα έτη 2018-2019. Δεύτερον, και για να περάσουμε στον ένα ευρύτερο πλαίσιο τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στη συμφωνία για την, στη συνθήκη μάλλον για την πώληση όπλων. Εδώ μιλάμε για ενιαία, γενικώ αποδεκτά ε, πρότυπα και προδιαγραφέ σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων. Τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2014 αυτή η συνθήκη και ω τώρα 130 χώρε το έχουν υπογράψει, 92 ε, είναι ε, χώρες που έχουν, οι ε, πλέον χώρες που έχουν υπογράψει. Βεβαίως ε, ορισμένες σημαντικές χώρες εξαγωγής όπλων, Ινδία, Πακιστάν, Ρωσία, Κίνα ε, δεν έχουν υπογράψει ή επικυρώσει αυτή τη συνθήκη. Όλες οι διπλωματικές δυνατότητες χρησιμοποιούνται για να ενθαρρύνουμε τις χώρες που έχουν κάνει βήματα προς τη συνθήκη αυτή να προσχωρήσουν και όποτε χρειαστεί το, το πρόγραμμα ε, ενίσχυσης και αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη διάθεσή τους. Είναι ε, καθήκον μας ε, εμείς να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε ό,τι αφορά την εξαγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης καθήκον μας να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε και άλλους παραγωγούς κατασκευαστές όπλων να εφαρμόσουν τα πρότυπα του ITT, της συνθήκης δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τις πολιτικές ομάδες. Συγγνώμη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τον κύριο Κέλαμ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μάσκας, ευχαριστώ τη συνάδελφο Βαλέρο για το ανοιχτό της πνεύμα, την ετοιμότητά της, τη δέσμευσή της απέναντι σε διαφορετικές ε, απόψεις. Καταρχήν είμαι ικανοποιημένο που η έκθεση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της κάθε χώρας να προβαίνει στην αυτοάμυνά της. Ότι μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα όπλα για την αυτοάμυνά της. Τα οχτώ κριτήρια τώρα. Είναι επίσης μια ισχυρή δέσμευση των χωρών μελών που μιλάει για έλεγχο των εξαγωγών προϊόντων της εθνικής εκάστοτε βιομηχανίας όπλων πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια αυτά και αρχές. Υπάρχουν βέβαια διάφορα ε, προβλήματα με την υλοποίηση της κοινή θέση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση και πιο σαφής. Πάντως το ΕΛΚ δεν βλέπει να χρειάζονται νέα επιπλέον κριτήρια ή επιπλέον δομές ε, ή κυρώσεις για να επιβληθούν. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την υλοποίηση της κοινέ μας θέσης. Και αυτό που χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο είναι ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά για τις άδειες που δίνονται, για τις εξαγωγές που γίνονται. Οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικούς τρόπους να συλλέγουν πληροφορίες. Οπότε πρέπει να είμαστε σε θέση τακτικά να ανταλλάσσουμε πληροφορίες κάθε φορά που μια κυβέρνηση αποφασίζει να δίνει την άδεια ή να αρνείται την άδεια για εξαγωγές όπλων. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια πλατφόρμα όπου να ανταλλάσσουμε τέτοιες πληροφορίες. Αλλά έτσι κι αλλιώς το θέμα μας ανησυχεί, είναι αλήθεια ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του μέσω μιας κοινή στρατηγικής των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσαμε χωριστές ψηφοφορίες για τους παραγράφους 29 και 34 με το ECR ελπίζουμε οι συνάδελφοι να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Παρακαλώ, Ινέ, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τις ευχαριστίες προς την εισηγήτρια και με την ικανοποίηση που εξέφρασε και ο προλαλής σας όσον αφορά τη συνεργασία μας με την κυρία Βαλέρο. Ήταν πολύ θετική. Και την ευχαριστώ επίσης γιατί συμπεριέλευε και κάποια καινοτόμα στοιχεία όπως είναι η δυνατότητα να υπάρξει κατάλογος με οντότητες ή με ιδιώτες τους οποίους υποψιαζόμαστε ότι εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο όπλων ενώ εμφανίζονται σαν εταίροι μας. Επίσης, τη δυνατότητα να ενσωματωθεί κάτι για την ασφάλεια απέναντι σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και αναφέρουμε και τις δυνατότητες απειλών σε εθνικά δίκτυα κλπ. Όλους αυτούς τους κινδύνους. Οπότε είναι καλό που έχουν συμπεριληφθεί γιατί πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ενημερώνουμε καλύτερα όσους εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ελέγχου. Τώρα θα έχουμε και το Brexit ε, στο μέλλον. Κάποια στιγμή δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πια μαζί μας. Οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα ελέγχου του τι γίνεται στο διεθνές εμπόριο όπλων. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια που έχει συμπεριλάβει και θέματα που έχουν να κάνουν με την κάλυψη και την προστασία των whistleblowers, των καταγγελόντων, οι οποίοι καταγγέλουν δικήσεις, ε, υπηρεσίες. Είναι καλό να υπάρχει αυτή η προστασία αυτών που καταγγέλουν παραβιάσεις στην κοινή θέση είναι καλό να γνωρίζουμε αυτές τις κακές πρακτικές, να υπάρχει δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας, οπότε αυτοί που τις καταγγέλουν πρέπει να προστατεύονται. Και είναι καλό επίσης να ταμείβονται και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τους καλούς κανόνες. Σωστά. Επίσης, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εκείνες των ΗΠΑ πρέπει να τις εντάξουμε στις δικές μας ρυθμίσεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Ευχαριστούμε κύριο Βανόρντεν. δύο λεπτά Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρέπει να θυμόμαστε βεβαίω ότι είναι ζωτικά σημεία και της εθνικής μας ασφάλειας αλλά και της οικονομικής μας ευημερίας ε, η παραγωγική κλάδη των, ε, των, της οπλικής βιομηχανίας. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό εσόδων από τις εξαγωγές όπλων και έχουμε πολύ, καλή, ε, πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο και στην παραγωγή αλλά και στις εξαγωγές όπλων. Και αυτό με τον όρο ότι δεν θα καταλήγουν σε λάθος χέρια είτε όπλα είτε, είτε τμήματά τους είτε σε, κράτη τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα είτε σε τρομοκράτες είτε σε άλλους εγκληματίες. Όλα αυτά έχουν εξασφαλιστεί από την νομοθεσία και η δική μου η πατρίδα του Ρωμανού Βασίλειου έχει στεναρή και στεναρό και αποτελεσματικό γενικό σύστημα ελέγχονται των εξαγών όπλων ανεξαρτήτως μάλιστα της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ε, σε σχέση με την έκθεση της κυρίας Βαλέρο καταγράφουμε κάποια σημαντικά σημεία Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απορρίψει κάθε υπενιγμό κυρώσεων εναντί κράτου μέλου που δεν τηρεί ενδεχομένω κοινή γνώμη. Επίσης, δεν βλέπουμε αυτή τη χρονική στιγμή με τι οικονομικές, δημοσιονομικές πιέσεις. Δεν υπάρχει ένα λόγος λοιπόν να, ε, να δαπανηθούν χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για ανάπτυξη δυναμικού και προσωπικού διαχείρισης των αδειών ή ελέγχου των αδειών. Βεβαίως και υπάρχει διεθνή συνθήκη και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μάστικας για την έμφαση και τον τόνο που έδωσε στην υπόθεση αυτή. Αλλά πρέπει να διαρωτηθούμε. Υπάρχει λόγος να ενισχυθούν οι δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει η ευρύτερη διεθνή κοινότητα που θα πρέπει να αναλάβει από πλευρά της δραστηριότητα γιατί δεν γίνεται πουθενά λόγος ε, για τις χώρες που παραβιάζουν τα διεθνή συστήματα για τις ε, πωλήσει όπλων και παραβιάζουν όλες τις συμφωνίες σε διάφορα μέρη της γης, όπως η Ρωσία, το Ιράκ, το Πακιστάν, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα. Σε αυτά τα κράτη θα πρέπει να εστιαστούμε. Είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν προσπογράψει την Συμφωνία για τα Όπλα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συμβαλόμενα μέρη της σχετικής συνθήκης. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, έχετε μπλε κάρτα, κύριε Βανόρντεν. Εκ μέρους της κυρία Σκότ, κατώ. Τη δέχεστε. Εξάπαντος, λέει ο κύριος Βανόρντεν. Παρακαλώ την ε, ερώτησή σας. Αυτή η συζήτηση για τις εξαγωγές όπλων έχει να κάνει με την μεγάλη έκθεση, διεθνή έκθεση όπλων στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή και ύστερα από την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορίου στην Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βανόρντο, θα συμφωνήσετε με την έκθεση της κυρίας Βαλέρου ε, που ζητάει να σταματήσουν οι πωλήσει όπλων Σαουδική Αραβία που τα χρησιμοποιεί για να σκοτώνει παιδιά στην Ιεμένη. Κύριο Βανόρντεν, ναι, είμαι βεβαίω ότι είχατε ετοιμάσει την ερώτηση σα πριν αρχίσω να μιλάω καν. Και πρέπει να πω ότι δεν μου αρέσει και ο τόνο με τον οποίο να απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε μένα. Βεβαίω και καταδικάζω πλήρως ε, τους, ε, τις δολοφονίες παιδιών ε, αλλά και κάθε αμάχο. Το να απαγορευτούν όμως οι εξαγωγές όπλων προς Σαουδική Αραβία, όχι δεν θα συμφωνήσω και πρέπει να πω ότι υπήρξε δράση της λεγόμενης εκστρατείας κατά το εμπορίου όπλων, γιατί από εκεί προερχόνται αυτές οι ιδέες, κατά της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έφτασε μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, το High Court, τον Ιούλιο του 2017 συγκεκριμένα ε, δόθη ετοιμιγορία υπέρ του Τη ε, της του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, δεν έχω το χρόνο να σας διαβάσω όλο το σκεπτικό της απόφασης, πολύ ευχαριστώ να τη διανύμω όμω. Και πάντως σημειώνει στην ετοιμιγορία ότι η απαγόρευση η απόφαση του Υπουργού ε, Εμπορίου ε, για τη μη απαγόρευση εξαγωγών όπλων προς τη Σαουδική Αραβία δεν ήταν ούτε παράλογη ούτε ακραία. Αυτά ως, το προς το κύριο σκεπτικό. Ευχαριστώ πολύ. Να να εκ μέρους της Άλντε. Ενάμιση λεπτό εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας παρακαλώ να μην μπερδεύουμε ε, την νόμιμη άμυνα όπου χρειάζεται όντως ε, άμυνα, να μην το ε, μπερδεύουμε με το εμπόριο. Τα 8 κριτήρια που υπάρχουν το 2008 πρέπει να ε, εφαρμοστούν, όχι να είναι απλά λόγια. Και η πραγματικότητα είναι η εμένη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βομβαρδίζονται με προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη. Made in Europe. Αυτό είναι ντροπή. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχιστεί επειδή το εμπόριο του αίματος πρέπει να συνεχίσει να ρέει για να υπάρχει η πραγματικότητα της άμυνάς μας. Η νόμιμη άμυνα δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να τηλερώνουμε με το αίμα άλλων. Έχουμε εγκρίνει αυτά τα οκτώ κριτήρια και πρέπει να τα διατηρήσουμε. Βεβαίω, ε, παραδείγματο χάρη υπάρχουν κυρώσει για περιπαραγωγή γάλακτο, έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσει λοιπόν όταν πολλούνται όπλα έξω από αυτά τα οκτώ κριτήρια και υπάρχουν χώρε οι οποίε στην πρώτη γραμμή των, εξαγωγών που παραβιάζουν τα οκτώ αυτά κριτήρια. Είτε λοιπόν σεβόμαστε αυτά που έχουμε ε, ε, αποφασίσει ή ας καταργήσουμε τα οκτώ κριτήρια. Ας είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε τίμοι. Πουλάμε σε όποιον αγοράζει. Διότι έχει σημασία μόνο το εμπόριο και όχι η ηθική. Αυτό είναι το βασικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόζινγκ εκ μέρου τη ΓΟΥ, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Ακούω να μιλάει ο κύριος Βανόρντεν και φαντάζομαι ότι όλα έχουν ε, διευθετηθεί κατά εξαιρετικό τρόπο αλλά είναι πολλές οι μελέτε που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και ο κύριος Νάρτ πολύ εύστοχα μιλάει για τα εγκλήματα στην Ιεμένη. Πρέπει λοιπόν πια αυτό, αυτή η παράνοια να βρει όρια. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε πρόοδο στον τομέα αυτών βεβαίως, αλλά πάνω απ' όλα, και αυτό το τονίζει η έκθεση, τα οκτώ κριτήρια ορίζουν ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορισμό δηλαδή των εξαγωγών και για τον κύριο Κέλαμ. Δεν πρόκειται καθόλου για νέα κριτήρια, κύριε Κέλαμ. Πρέπει να ε, διαπιστώσουμε ωστόσο, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, για να μην πω όλα, παραβιάζουν παγίω αυτέ τι προδιαγραφέ. Η Γερμανία, γιατί δεν μιλάμε σήμερα για Ρωσία. Η Γερμανία, παραδείγματι, με βάση τι μελέτε, ε, το 2015 και μόνο έκανε 4, έδωσε 4.000 εξαγωγικέ άδειε σε 27 διαφορετικέ χώρε, οι οποίε ε, θα, θα υπάγονται στα κριτήρια απαγόρευση. Επομένως ε, και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Χρειάζονται τρία βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε συγκεκριμένε προδιαγραφές ε, και τήρησή τους. Χρειάζεται ενιαίο και επιτέλους ε, και επιτέλους ταχύτερη καταγραφή και υποβολή των εκθέσεων από τα κράτη-μέλη και επίσης ανεξάρτητη επαλήτευση από ανεξάρτητες πλευρές αλλά και μηχανισμοί κυρώσεων κατά των κρατών που επιμένουν στην παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού και επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται με την εξαγωγή των όπλων η επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με τις εμπόλεμες συγκρούσεις όλο τον κόσμο. Η κυρία Λούνατσεκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι στην συζήτηση βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ε, ποιοι είναι οι λόγοι των μεταναστευτικών ροών που οδηγούν πολλούς ανθρώπους στα σύνορα των κρατών μας. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια οι οικονομικές συνθήκες αλλά και οι εξαγωγές των όπλων και κυρία Βαλερό νομίζω αξίζει συγχαρητηρίων και ευχαριστειών για την εξαιρετική της έκθεση γιατί ορίζει, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά δεσμευτικέ θέσει του 2007 και δεν θα πρέπει σε κράτη τα οποία ε, βρίσκονται σε πολέμη κατάσταση ή παραβιάζουν τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα να εξάγονται όπλα. Πρέπει να απαγορεύεται λοιπόν η εξαγωγή όπλων και αυτό πιστεύω ότι πρέπει αμέσω να εφαρμοστεί σε σχέση με την ε, Σαουδική Αραβία η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με την ε, Ιεμένη και αυτό ήδη έχει αναφερθεί από του συναδέλφου, Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταδικαστεί. Επίσης είναι ότι εξάγονται ακόμη ε, όπλα προς τη Σαουδική Αραβία. Η Αυστρία ίδια πέρσι 30.000 μικρά όπλα εξήγε. Θα πρέπει λοιπόν προς την κυρία Μογκερίνη να απευθύνουμε το μήνυμα για ένα εμπάργκο όπλων ε, έναντι της Σαουδικής Αραβίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η FDD, Κάρβερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εξαγωγή όπλων θα πρέπει ε, να εξαρτάται από ανεξάρτητες και πραγματικά κυρίαρχες κυβερνήσεις. Σε πολλούς τομείς ε, πολιτικής της δικής μου κυβέρνησης μπορεί να μην υπάρχει αυτό. Ε, θεωρώ πραγματικά πρέπει να εξαρτάται και να βρίσκεται πλήρως στα χέρια των ψηφοφόρων της κάθε χώρας. Και γιατί ένα τέτοιο σημαντικό στοιχείο πάντα λαμβάνεται υπόψη και κατά μία εκλογική, προεκλογική εκστρατεία. Λέτε ότι μετά τον Brexit θα πρέπει να ξεκολουθείτε να συνδέετε από την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ απορρίπτω ε, εντονώς ε, αυτή την ε, στάση μέσω ε, του μελλοντικού... Υπάρχει μάλλον δημοσιεύτηκε σήμερα ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο είναι μάλλον ασαφές όμως και δεν είναι πλήρες. Για να κερδίσουμε και πάλι πλήρως την ανεξαρτησία μας σε αυτόν τον τομέα, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποσυρθεί από την κοινή ε, στρατιωτική δομή και όπου δει να αξιοποιεί το ΝΑΤΟ. Αυτό ψήφισε, ε, ψήφισαν οι Βρετανοί όταν ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι. Ευχαριστώ κύριο Σαφχάουζερ, παρακαλώ, από το ΙΕΝΕΦ για ένα λεπτό. exportations d'armement des États membres. Οι εξαγωγέ όπλων των κρατομελών, ενώ η χρήση ε, και οι κανόνε που του διέπουν ήδη περιορίζουν την ελευθερία στα κράτη μα. Το έχουμε δει με, τους, ε, με τα Μιστράλ, που παρά τις υποσχέσεις ε, η Γαλλία είδατε τι στάση κράτησε. Και έχουμε παρακολουθήσει τις συστάσεις. Ωστόσο, όταν τα δυτικά όπλα πρέπει να φτάσουν στα χέρια των ε, ομάδων νεοναζί όπως στην Ουκρανία ή των τζιχαντιστών όπως στη Συρία ή στη Μέση Ανατολή που έχει μια ιδιαίτερη ε, θέαση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τότε υπάρχει δυνατότητα και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ορισμένες χώρες δεν μπορούμε να υποτάξουμε την ε, αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της Γαλλίας ε, στο εξωτερικό. Έχει σχέση με την εθνική μας κυριαρχία, έχει έρθει η ώρα να φύγει η Γαλλία από αυτή την Ευρώπη. Ο κύριος Γκάλερ για 1,5 λεπτό είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να καλωσορίσω τον κύριο Μάσικα ε, και να τον ευχαριστήσω για την εισαγωγική του ομιλία. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση κάθε χρόνο, διότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την εξωτερική μας πολιτική και θα έπρεπε, πιστεύω, τουλάχιστον καταρχάς να αναγνωρίσουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη περιφέρεια στον κόσμο που έχει έναν τόσο απαιτητικό κατάλογο κριτηρίων για την εξαγωγή ή μη εξαγωγή όπλων. Έναν κατάλογο ε, που πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει μιμητές σε άλλες χώρες του κόσμου. Βέβαια, είναι και ρεαλιστικό από την άλλη πλευρά να ε, να γνωρίζουμε ότι δεν θα υπήρχε σε αυτή η κοινή θέση του Συμβουλίου αν δεν ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν με βάση αυτά τα κριτήρια για το τι θα κάνουν ή αν δεν ασχολούνται με αυτό το καθήκον πιο σοβαρά τα κράτη-μέλη. Φαίνεται λοιπόν ότι στο πλαίσιο των ε, αρμοδίων ε, ομάδων εργασίας του Συμβουλίου γίνεται σε τακτά διαστήματα συζήτηση για το πώς έχει κατάσταση διάφορες ε, πόλεμες ζώνες. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν το αποτέλεσμα τέτοιων συζητήσεων να είναι ότι ε, θα υιοθετούσαμε την ίδια ε, κοινή άποψη για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο. και οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη να κάνουν αυτή τη συζήτηση και όχι άλλοι. Ευχαριστώ. Κύριος Πίτσουλα έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση ορθώς τονίζει ότι για τα κράτη είναι θεμητό να για τους. Μην ξεχνούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να υποβάλλονται οι σωστές εκθέσεις και αναφορές και επίσης θα πρέπει νομίμως να ενεργούν οι εταιρείες που παράγουν τα όπλα. Έχουμε σχεδόν 100 δις αδειών που εκτείνονται για εξαγωγή όπλων. Αυτό είναι τεράστιο νούμερο. Χρειάζεται διαφάνεια. Χρειάζεται να ξέρουμε πού καταλήγουν αυτά τα όπλα. Η διεθνή κοινότητα συχνά αντιδρά πολύ αργά. Αφού έχουν αρχίσει κάποιες σύγκρουσεις, χρειάζονται κριτήρια ελέγχου των εξαγωγών. Να μην έχουμε κατάτμιση των πόρων, μην έχουμε επικάλυψη αυτών και να σταματήσει ε, αυτή η διεύρυνση και επέκταση των ε, εξαγωγών. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την άμυνα, ε, με την, με Ένωση της Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Τόμασιτς ε, αυτές οι εξαγωγέ προς τρίτες χώρες πολλές φορές καταλήγουν στα λάθος χέρια, οπότε έχουμε διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Έχουμε καταπάτηση των δικαιωμάτων. Έτσι κι αλλιώς ο πόλεμος είναι κάτι το καταστροφικό. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος δείχνει το χειρότερο εαυτό του αυτό, οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε να μην, πώς θα εκμεταλλεύονται αυτοί οι πολιτές όλων των πόλεμων, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιον κρίκο σαν λυσίδα μπορούμε να ελέγξουμε σαν λυσίδα αυτού του εμπορίου όπλων. Πως να μην σκοτώνεται κόσμος από αυτά τα όπλα. Προσοχή μπέσει στο κενό η προσπάθεια της υπάρξης εκπροσώπου. Ε, προσπαθεί κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν γίνεται τίποτα. Λέγεται ε, όμως νομίζω ότι δεν θα πρέπει τελικά να στηρίζουμε τους ε, μεγάλους κατασκευαστές όπλων. Ένα λεπτό, Ένα λεπτό. Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσπο. Μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθε, το Amnesty να λέει ότι κάθε ε, χρόνο 500.000 άνθρωποι σκοτώνται από πυροβόλα, όπλα και πολλές, πολλά εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι είναι πληγμένοι μέσα σε εμπόλεμες συγκρούσει και λόγω της αλόγης της εμπορίας όπλων. Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει σχολεία και άλλε ε, δομέ στην Ιεμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που εκπαιδεύονται και φέρουν σε πέρα στρατιωτικές αποστολέ και επιχειρήσει στην Ιεμένη και σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, αυτό που ζητούμε εδώ είναι όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από την Ισπανική κυβέρνηση συγκεκριμένα και από το Βασιλικό Οίκο να ε, ξαναδεί τι στρατιωτικέ και επιχειρηματικέ σχέσει με χώρε όπω είναι το, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα ποτέ δεν μπορούν να, να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική ούτε να είναι πιο πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πολύ θετικά στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή των διεθνών συνθήκων, με τα σεβασμό των δικαιωμάτων και με τη διαφάνεια. Καταλαβαίνουμε ότι το βασικό δεν είναι μόνο να υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση, αλλά να αναλάβουμε δέσμευση εδώ να μην μείνει κενό γράμμα. Ευχαριστώ. Μπούχνερ τώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το ο Κοινοβούλιο σήμερα ξεκάθαρα μίλησε για τις εξαγωγές όπλων σε εμπόλεμες περιοχές. Όμως η Γερμανία, η πατρίδα μου, δυστυχώς είναι ένας από τους βασικούς εξαγωγείς όπλων στον κόσμο σε περιοχές όπου σοβούν συγκρούσεις. 24 ε, ε, Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα νέο καγκελάριο, είτε την κυρία Μέρκελ τον κύριο Σούλτ. Τα ίδια θα γίνουν όμω, όποιο και αν εκλεγεί. Μέρκελ, Γκάμπριελ, Σούλτ πρέπει να ε, ε, ξέρουμε ότι παρουσιάζονται μένως οι ήρωες και οι σωτήρες ε, των μεταναστών, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι χώρες ε, όπως Κατάρ, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία τις προμηθεύουν με όπλα. Οι γερμανικές εξαγωγές ε, χρησιμοποιούνται τα όπλα αυτά δηλαδή για ε, την καταπίεση των δικαιωμάτων. Το ίδιο γίνεται στην Τουρκία που χρησιμοποιούνται τα γερμανικά όπλα κατά των Κούρκων. Το ίδιο κάνει η Σαουδική Αραβία κατά της Ιεμένης. Η Αίγυπτος βομβαρδίζει το δικό της τον πληθυσμό από ό,τι ε, φαίνεται και από ό,τι λένε για να ε, αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες. Αλλά είναι πραγματικά απαράδεκτο ε, να θέλουμε να καταργήσουμε και να εκριζώσουμε τους λόγους της μετανάστευσης και δεχόμαστε τους μετανάστες εδώ ενώ έχουμε δώσει όπλα για την εξόντωση αυτών των ανθρώπων στις χώρες τους. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Ένα λεπτό. Πέρασε πάνω από 1,5 χρόνος από το που συζητήσαμε το προηγούμενο θέμα που αφορούσε την κοινή θέση για τις εξαγωγές των όπλων. Λίγα όμως ε, αλλάξανε και όλη αυτή η business συνεχίστηκε τα κράτη-μέλη και βλέπουμε ότι ε, ε, Αίγυπτο, Σαουδιά Αραβία και Τουρκία είναι οι προορισμοί των εξαγωγών μας χώρες που δεν είναι και τόσο δημοκρατικές να πούμε το λιγότερο. Θα πρέπει να υπάρχει εκείνο το εμπάργο που είχαμε πει το 16 στο Ριάντ ε, έγινε αυτό που υπήρχε το εμπάργο της παραβίαση της ε, απόφασης του εμπάργου από 157 εκατομμύρια η χώρα μου εξέγει όπλα 427 ε, μέσα σε ένα χρόνο οπότε και συνεχίζουν οι άμαχοι και τα παιδιά να σκοτώνουν με αυτά τα όπλα τα δικά μας χέρια είναι λερωμένα. Δεν έχουμε έλεγχο, καμία εκκύρωση, απλώς υποκριτικά κινούμεθα με επίφαση ε, Ευχαριστούμε την ε, κυρία Βαλέρα. Το 2012 πήραμε την, το, το, το βραδείο για την ειρήνη. Ας ότι το αξίζαμε. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εθνική άμυνα είναι μια εθνική αρμοδιότητα και έτσι πρέπει να παραμείνει. Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να ε, αποκτήσει ε, στρατιωτική τεχνολογία για την άμυνά του και έχει το δικαίωμα να εξάγει όπλα. Υπάρχουν όμως ε, διάφορα παράνομα ε, σχέδια επιστροφής αυτών των όπλων, ε, ακόμα και μέσω των δημοκρατικών οργανώσεων. Στηρίζω λοιπόν την έκθεση Βαλέρο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Επίσης συμφωνώ σε ό,τι αφορά το εμπάργκο στη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη όμως η έκθεση Βαλερό ε, πραγματικά θεωρώ ότι αποτελεί σκάνδαλο όταν θέλει να δώσει στην Ένωση το δικαίωμα να διοδοτεί ή όχι τι χώρε μέλη για να εξάγουν τα όπλα. Αυτό είναι θέμα ε, εθνικής κυριαρχίας, γι' αυτό και θα καταψηφίσω την έκθεση. Κυρία Αλιομαρή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλούμε για την εθνική άμυνα, ε, όταν πρόκειται για την εξαγωγή όπλων δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Σήμερα βλέπουμε ότι οι χώρες ε, μεγάλη εξαγωγή ε, όπλων, πιο συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκές χώρες, στηρίζουν και σέβονται τους πολύ αυστηρούς κανόνες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Η Γαλλία, για παράδειγμα, ε, έχει ακόμα πιο αυστηρά πρότυπα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Πρέπει επίσης όταν μιλούμε για τέτοια ζητήματα να επενθυμίζουμε την ε, σύγκληση των συμφερόντων τελικά των χωρών έναντι της τρομοκρατίας, έναντι της ε, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου απέναντι ε, στην αποσταθεροποίηση σε ε, αρκετές χώρες. Οπότε υπάρχουν ε, χώρες και περιοχές όπου έχουμε τοπικές συγκρούσεις, αλλά ένα και περισσότερο διεθνοποιούνται αυτές. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα αλληλεγγύης εδώ και δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα σε αυτές τις χώρες να αμυνθούν. Τώρα αυτό που λένε για την απαγόρευση των εξαγωγή των όπλων είναι μια πρόταση καθαρά ιδεολογική. Θέλουμε να στερήσουμε το δικαίωμα στα, σε ένα κράτο δικαίου να ε, αμυνθεί, να περισσεύει αυτό εαυτό του. Είναι μια αφέλεια. Ε, αφέλεια να θεωρούμε ότι μπορούμε να στερήσουμε αυτό το δικαίωμα στου πολίτε μας να αμυνθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα το ε, δικαίωμα στην εξαγωγή των όπλων και ότι αυτό που θα πρέπει να γίνεται βάσει κανόνων, σαφώς και είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Όμως ε, η τυφλή και συνολική απαγόρευση ε, είναι αρνητική. Υπάρχει γαλάζια κάρτα, αν τη δέχεστε. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κυρία Λιωμαρή. Λέτε ότι είναι ειρηνική αυτή η έκθεση και ότι δεν μπορούμε να απαγορεύουμε τις εξαγωγές όπλων. Η κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων αποφασίστηκε από τις κυβερνήσεις, από τα κράτη-μέλη, άρα και από τη Γαλλία. Και υπάρχουν αυτά τα οκτώ κριτήρια ε, με βάση τα οποία επιλέγεται σε ποιες χώρες εξάγονται όπλα. Η Σαουδική Αραβία είναι σε πόλεμο με την Ιεμένη. Είναι ένα κριτήριο αυτό. Επίσης βομβαρδίζονται μη στρατιωτικοί στόχοι. Το βλέπουμε. Ε, βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές. Υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τραυματίες και νεκροί από όπλα τα οποία έχουν αγοράσει από τη Γαλλία, τη Γερμανία, ίσως από τη Μεγαλτένια και άλλες χώρες. Αυτό θεωρείτε ότι είναι λογικό και να μας λέτε εδώ αυτές τις ανοησίες τις ειρηνευτικές όταν ε, ε, κινδυνεύει τόσος κόσμος από αυτά τα όπλα. Εσείς κυρία μου έχετε το λόγο, κυρία Λιωμάκη, για να απαντήσει. Χωρίς μικρόφωνο. Ξέρω τι είναι ο πόλεμο και ω υπουργό Άμυνα ε, πήγα σε αυτέ τι εμπόλεμε ζώνε και είδα πραγματικά τι ήταν ο πόλεμο. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα γνωρίζω. Στο ερώτημά σα, ε, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά τα κριτήρια. Πράγματι έχουν θεσπίσει τέτοια κριτήρια αυτέ οι χώρε και το είπα ε, ότι οι Ευρωπαϊκέ χώρε έχουν θεσπίσει τα κριτήρια και σα είπα επίση ότι η Γαλλία είναι αυτή που έχει τα πλέον αυστηρά κριτήρια σε ολόκληρο τον κόσμο σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ όπλων. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον για τη Σαουδική Αραβία. Μίλησατε πολύ για τη Σαουδική Αραβία. Εγώ προεδρεύω της ε, αντιπροσωπείας ε, με τις ε, χώρες του περσικού κόλπου. Αν θέλετε να μιλήσουμε τότε, να μιλήσουμε και για το Ιράν και για εκείνου που δημιουργούν εξίσου μεγάλες καταστροφές για τον πληθυσμό που δεν είναι η Σαουδική Αραβία, είναι άλλε χώρε. Και να σας υπενθυμίσω ότι ο συνασπισμός των χωρών του Περσικού έχει ε, παρέμβει ε, κατόπιν αιτήματος ε, του, της ημενικής κοινότητας. Εσείς λέτε τελικά στηρίζετε τους ε, αντιστασιακούς έναντι των, της ε, νόμιμης κυβέρνησης. Ναι, ναι. Ένα λεπτό κύριε Γκόμες. Συμφωνώ με όσο είπε η κυρία Λούνατσεκ στην κυρία Λία και υπενθυμίζω ότι η Γαλλική Προεδρία προέταξε και διαμόρφωσε αυτή την κοινή θέση. Και τώρα ήθελα να πω σε σχέση με την συγκήτρια ότι είναι πρόβλημα οι εξαγωγές γιατί και η Γαλλία μεταξύ άλλων κρατών δεν τηρούν τα κριτήρια εξαγωγής. Το Φεβρουάριο του 2016 με τις εξαγωγές προς Σαουδική Αραβία ζητήσαμε εμπάργο. Ήταν εγκληματικός ο πόλεμος κατά τις Ιεμένες. Πολύθηκαν τα όπλα χωρίς να εξεταστεί το καθεστώς της χώρας του εισαγωγής. Όλα αυτά είναι απειλή προς την ασφάλεια όλου του κόσμου και της Ευρώπης. Με το εμπόριο ξαναμπαίνουν τα όπλα στην Ευρώπη. Πάνε στους τρομοκράτες και στη Γαλλία. Άρα χρειάζεται μια εξάρτητη αργή, αρχή για έλεγχο, για κοινοποίηση για κυρώσει. Θα πρέπει να γίνεται και έλεγχος μετά τις εξαγωγές, ούτω ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω εμπορία αυτών των όπλων. Και θα πρέπει και μετά τον Brexit να δεσμεύεται η Ευρώπη από αυτές τις κοινέ θέσεις. Να Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε ο κύριος Φιέλνερ, για το θέμα αυτό. Εύκολα κανείς μπορεί να λαϊκίσει. Τα όπλα είναι κάτι το φρικτό γιατί σκοτώνουν τους ανθρώπους, άρα να απαγορεύσουμε εμπόριο, εξαγωγές κλπ. Όμως, είναι θέμα πολιτικής ασφαλείας και άμυνας εξαγωγής τεχνητικού υλικού. Και τα πράγματα εκεί δεν είναι άσπρο και μαύρο, απλά. Ποιος, ποια εταιρεία πουλάει σε ποιον και πότε, αυτό θα πρέπει να κρίνεται περιπτωσιολογικά. Αφήστε που τα πράγματα μέσα στον χρόνο μεταβάλλονται. Άρα το θέμα είναι ποιος θα τα αποφασίσει για το τι πρέπει να γίνει. Στην Σουηδία πάρα πολύ λίγοι πολιτικοί θα έλεγαν ότι χρειάζεται να αλλάξει το καθεστώς Εμεί οι Σουηδοί θέλουμε να αποφασίζουμε για τη Σουηδική άμυνα, για τα Σουηδικά όπλα, για τη Σουηδική πολιτική ασφάλεια. Και η αριστερά, πράσινη και κόκκινη λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή θέση, θα πρέπει να υπάρχουν κοινέ κυρώσει. Μα αυτό είναι διακυβερνητικό. Αυτό μα αφαιρεί κυριαρχία. Δεν είναι επικουρικότητα και η επικουρικότητα δεν είναι κάτι που σβήνουμε και ξανανάβουμε ανάλογα με το τι αρέσει στους ψηφοφόρους. Άρα θα πρέπει να ε, αποφύγουμε το λάθος, να έχουμε αυτές τις κοινές θέσεις για την εξαγωγή. Κύριε Φιέλνερ, υπάρχει μια γαλάζια μπλε τέλο πάντων κάρτα για εσάς. Την αποδέχεστε, κύριε Φιέλνερ, μάλιστα λέει και η κυρία Βαλέρο, η συγγήτρια, θα κάνει την επερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Φιέλνερ. Η κοινή θέση είναι το ελάχιστο. Δεν είμαι κανείς για το δικαίωμα της Σουηδίας να αποφασίζει. Και ξέρετε πολύ καλά, όπως ξέρω και εγώ, ότι ισχύει στην ε, Σουηδία. Υπάρχει μια κοινή πολιτική και το δικό σας κόμμα συμμετέχει, το δικό μου κόμμα. Δεν λέω πουθενά στην έκθεση τίποτα το αντίθετο. Η απάντησή κύριε Φιέλνε. Ευχαριστώ. Δεν είπατε όμως ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ τη τωρινή κοινή θέση και αυτού το οποίο εσεί προτείνετε. Το θέμα είναι οι κυρώσει. Το πρόβλημα είπαμε μεταβάλλονται στον χρόνο. Έχει την ευκαιρία τώρα να θεσπίσει κάποιε κυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αν κάποια χώρα διαφωνεί, τότε η ρύθμιση αυτή είναι διεθνή είναι διακυβερνητική. Είμαι βέβαιο ότι θα περάσει με ευρεία πλειοψηφία η έκθεση και εσείς θα πάρετε πολλούς επένους αλλά δεν νομίζω ότι το θέμα των κυρώσεων ποτέ θα υλοποιηθεί διότι τα κράτη και εγώ θεωρούν ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και διεθνείς κυρώσεις δεν θα περάσουν. Σωράγια. Έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Μποντίλ Βαλέρο για την ε, έκθεση αυτή. Είμαι πρόσωπο τη φεμινιστική πρωτοβουλία ε, και της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας ε, και εμείς πασιφιστές δυσκολευόμαστε να ψηφίσουμε υπέρ της εξαγωγής όπλων υπό οποιαδήποτε μορφή. Πάντως σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος των εξαγωγών όπλων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είδαμε ότι το εμπόριο, οι εξαγωγές όπλων ανθούν, λέει ο Economist. Δεν μπορούμε να το ε, μην λαμβάνει υπόψη και την ιστορική απόφαση του ΙΕΣ 17 για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων. Και η, το ειρηνευτικό φεμινιστικό κίνημα ε, για χρόνια αγωνιζόταν και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να επιβληθεί η απαγόρευση αυτή. Λέγανε ε, στους ακτιβιστές δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Να όμως που έκαναν λάθος. Ε, άρα μπορούμε να καταργήσουμε τα όπλα και έτσι μόνο θα αλλάξουμε τον ε, κόσμο με, μια φεμινιστική, με ένα φεμινιστικό όραμα για τη δημιουργία ενός ειρηνικού κόσμου χωρίς όπλα και με το διάλογο μόνο ως όπλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παρνιό έχει το λόγο. Σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχει αταξία, κίνδυνος, ε, στάθεια, είναι σαφές ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ε, την Ευρώπη της άμυνας. Χθε αυτό ήταν μια πραγματικότητα και σήμερα γίνεται αναγκαιότητα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια με βάση και τις αξίες μας, ε, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη υπευθυνότητα για τη δημιουργία αυτή τη αμυντική Ευρώπη Έχουν γίνει γιγαντιαία βήματα, άλματα το τελευταίο καιρό και πρέπει να τα στηρίξει το Κοινοβούλιο. Εμπιστοσύνη ταυτόχρονα όμω, γιατί σε ένα κράτο δικαίου θα πρέπει να γίνεται απόδοση λογαριασμών και αυτή είναι η πρόκληση τη έκθεση, Βαλέρο, που πολύ σωστά ζητάει να υπάρχει έλεγχο των εξαγωγών όπλων για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στον τομέα αυτό. Υπευθυνότητα λοιπόν σε μια Ευρώπη τη Άμυνας που θα μας προστατεύει, εμπιστοσύνη, των συμπολιτών μας στις δράσεις μας για την συλλογική ασφάλεια. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μήνυμα που στέλνουμε σήμερα. Κύριε Σκοφεράτη, έχετε εσείς τον λόγο. Για ένα λεπτό, Σέρτζο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι πεπισμένο ότι χρειάζεται νέε, πιο αυστηρές διατάξεις η Ευρώπη που να ρυθμίζουν τον έλεγχο των εξαγωγών των όπλων. Αυτό το πλαίσιο που προτείνεται είναι ανησυχητικό. Ε, είδατε τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτα-πρώτα αναφέρθηκε και σήμερα ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές ε, των 28. Το δεύτερο πρώτο προσέξουμε γιατί δεν έχει προβληθεί συστηματικά και με αυξανόμενο ρυθμό καταπατούνται τα κριτήρια που θα έπρεπε να διέπουν τις εξαγωγές, το εμπόριο τέλο πάντων προς τις χώρες που θέλουν να αγοράσουν τους ε, Ευρωπαίους χωρί χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις, τότε θα συνεχίσουμε να κηρύσουμε την ειρήνη και πολλές φορές έστω ε, τυχώς να το ξέρουμε αλλά συνεχίζουμε να έχουμε την ευθύνη μας να τροφοδούμε τον πόλεμο άρα θα πρέπει να κάνουμε αυτά που είπε η εισηγήτρια Ευχαριστούμε κύριε Φροντζούλικα, θα κλείσετε εσείς τη συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνεπή και λογική υλοποίηση της κοινή θέσης. Πολύ βασική για την αξιοπιστία της ε, Ένωσης. Μια που είμαστε διεθν, παίκτες διεθνούς κοινής, να γίνει έλεγχος των όπλων και των εξαγωγών να είναι αποτελεσματικό ο έλεγχο με διαφάνεια αποδεκτό από όλου, άρα τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τη δεσμευτικότητα τη κοινή θέση και θα πρέπει να πληρούν τι προποθέσει που έχουν τεθεί. Χρειάζεται αυστηρή εφαρμογή των κοινών κριτηρίων, περισσότερη διαφάνεια στο σύστημα εξαγωγών, ιδίω να σκεφτούμε τα τελευταία στοιχεία που λένε ότι Μέχρι το 2016 είχαμε αύξηση της τάξης του 26-27% των εξαγωγών. Άρα να θεσπιστεί αυστηρός μηχανισμός κυρώσεων για τα κράτη-μέλη που δεν θα υλοποιήσουν την κοινή θέση. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι και τώρα αρχίζει το κατσιδιά με τον κύριο Λίτσα. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Κύριε Συγήτρια, από το 2008 έχουμε τα 8 κριτήρια για την εξαγωγή όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε πρόοδο στη διαδικασία για τις εξαγωγή όπλων και δεν τα τήρουν αυτά τα κριτήρια όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώ ε, γι' αυτό λοιπόν στηρίζω την πρόταση για επιβολή κυρώσεων σε όσα κράτη δεν τηρούν αυτά τα κριτήρια. Υπάρχει δε η επανειλημμένη απέτηση ε, για εμπάργκο ε, απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να έχουμε μια συνεκτική επιτέλους εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά την εξαγωγή όπλων και τεχνολογιών. Ε, και ε, ο Μάρτιν Σούλτς ε, τα λέει και λέει ότι αν έχουμε κράτη-μέλη να δίνουν πόπλα σε χώρες που δεν θα έπρεπε αυτό θα βρει μιμητές και σε άλλες χώρες και θα το κάνουν όλο και περισσότεροι. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη το ζητεί και σε ό,τι αφορά την απαγόρευση μικρών όπλων και σε ό,τι αφορά την μείωση των εξαγών. Το ζητά το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα πρόγραμμα. Θέλουμε μια κοινή πολιτική για όλη την Ευρώπη. Σε Ευχαριστώ πολύ. Κυρία να έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση δείχνει πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. είναι τεράστιες εξαγωγέ ε, όπλων. Το 86% φτάνει στη Μέση Ανατολή. Πολύ σωστά αναφέρεται ότι ορισμένα κράτη-μέλη συνάπτουν ε, στρατηγικές ε, συνεργασίες και συμμαχίες με χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση. Όμως ελπίζω να μην ε, πιστεύετε αυτό που έλεγε ο Μπούς κάποια στιγμή ότι όσο περισσότερο στρατιώτε έχουμε τόσο περισσότερη ειρήνη θα υπάρχει. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγέα όπλων στον κόσμο. Αυτό κοστίσει ζωές. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, ως γνωστόν, οι αμυντικές βιομηχανίες... συμβάλλουν σημαντικά στη θωράκιση των εθνικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και στο ποσοστό ΑΕΠ κάθε κράτους μέλου. Όμω υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό και ατιμορρησία εταιρεών μεγάλων κρατών εξαγωγέων οπλισμού οι οποίε εμπλέκονται σε σκάνδαλα και παράνομε χρηματοδοτήσει με σκοπό την εξασφάλιση αντίστοιχων συμβολέων. η εφαρμογή ενωσιακού πεδίου εξαγωγή όπλων δεν θα δώσει λύσει προ αυτή την κατεύθυνση αλλά θα δημιουργήσει εμπόδια στι διασυνοριακέ πωλήσει αμυντικού οπλισμού και τι πωλήσει προ τρίτε χώρε. η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία ω ζωτικό παράγοντα για την αξιοπιστία τη εκολαπτώμενη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία λόγω της ύπαρξης διαφορετικών αμυντικών αντικειμενικών σκοπών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και της ταυτόχρονης ανυπαρξίας κοινών αμυντικών προσανατολισμών απόδειξη η παντελής αποσία της ένωσης στην έμπρακτη αντιμετώπιση της επιθετικότητας της τουρκίας έναντι της ελλάδος και της κυπριακής δημοκρατίας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε πολύ εδώ ε, που είμαστε πολλοί πασιφιστές, όμως δεν πρέπει να είμαστε και αφελείς. Γι' αυτό και εγώ χαιρετίζω αυτή την ισορπημένη έκθεση κυρίας Βαλέρο επιμένει σε κάποια στοιχεία τα οποία είναι ουσιαστικά και η άμυνα αλλά και η βιομηχανία των όπλων και δεν πρέπει να μας τα ούτε σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ούτω καθεξής έχουν ε, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές βιομηχανίες όπλων. Όμως αυτό που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτή την έκθεση είναι τα κριτήρια που θέλει να προωθήσει ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εισαγωγή και σε εθνικό επίπεδο και διεθνώ ε, και η αρχή τη προφύλαξη. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί υπάρχουν ε, όπλα και τεχνολογίες που ε, κινούνται προς χώρες που δεν είναι υπέρ τη ειρήνης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και κανόνε, Λογοδοσία λοιπόν και διαφάνεια και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό. Ευχαριστούμε. Κυρία Μωράη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ουγγαρία, η χώρα μου, εδώ και χρόνια λέει ότι ε, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης πρέπει να εξετάσουμε την ουσία του προβλήματος. Οι ένοπλες συγκρούσεις δημιουργούν τις μεταναστευτικές ροές. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε ποιος ευθύνεται, όχι η Ουγγαρία δεν φταίμε εμείς. Ποιανού ήταν αυτή η εξαιρετική ιδέα ε, της ανατροπής ε, του καθεστώτος Ασάντ στην Συρία και της παροχής όπλων ε, σε συγκεκριμένες ομάδες που αποδείχθηκαν τελικά τρομοκράτες. Ε, μάλλον αυτοί που ε, κέρδισαν πολλά από όλη αυτή την ιστορία. Αυτοί α υποδεχθούν του πρόσφυγες λοιπόν. Ποια ήταν αυτή η εξαιρετική ιδέα ε, ότι έχουν όπλα μαζική καταστροφή στο Ιράκ και ότι πρέπει να γίνει πόλεμο. Ποιο ωφελήθηκε από όλη αυτή την κατάσταση. Εκείνοι θα πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη λοιπόν ποιοι θεώρησαν ότι θα πρέπει να ανατραπεί το καθεστώς Καντάφη στη Λιβύη και ποιο θα μας σταματήσει όλες αυτές τις μεταναστευτικές ροές από την υποσαχάρια Αφρική. Είναι θέμα ευθύνη λοιπόν. Κύριε Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα φεστιβάλ, ένα παζάρι στα Ντόκλανς του Λονδίνου που αφορά όπλα και συναφή. Έχουμε πάνω από 1500 εκθέτες εκεί και έχουν για ελεύθερους σκοπευτές όπλα μέχρι ε, τάγκ, μέχρι πυράβλους κατά σκαφών και έχουμε επομένως εδώ χώρες που είναι οι πελάτες γιατί είναι βρίσκονται σε πόλεμο, είτε θέλουν να κάνουν καταστολή και έχουμε διάφορες ε, οργανώσεις που ε, υποστηρίζουν ε, αυτές τις κινήσεις αλλά το κάνουν αυτό κρυφά και έτσι οι έμποροι των όπλων κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να περιορίζονται από τους κανόνες και ουσιαστικά τη, την ύφη την πληρώνουν από την τσέπη τους. Δηλαδή οι Βρετανοί φορολογούμενοι συμφωνώ με όλους όσους είπαν ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Ο κύριος Καπούτο τελευταίος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 12 μέχρι το 16 το ποσό των όπλων ε, αυξήθηκε όσον αφορά τις εξαγωγές και ε, ε, μια πενταετία με τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του ψυχρού πολέμου και έχουμε επίσης εμπορίο προς χώρες που χαρακτηρίζονται προβληματικές. Έχουμε όμως την κοινή θέση και ιδίως προς Μέση Ανατολή έγινε εμπόριο. Επομένω, έχουν αλλάξει τα, τα πράγματα, έχουν γίνει πιο ασταθεί. Συνεχής είναι οι εξελίξεις. Θέλουμε αυτά τα νέα κριτήρια στην κοινή θέση να λαμβάνεται υπόψη ε, ο κίνδυνος που υπάρχει και το ότι μπορεί τα όπλα να εκτραπούν όσον αφορά για να ξαναγυρίσουν. Θα έχουμε συμφέρον το κάνουμε αυτό. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με μεταξύ ΚΟΑΡΜ και ε, των άλλων φορέων. Οπότε χρειάζεται να δούμε ποιε είναι οι χώρε προορισμοί και ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες τεχνολογίες που εμεί στην Ευρώπη παράγουμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Κύριε Μάσικα, ε, ο λόγο ξανά σε εσά. για τη συνέχεια της συζήτησης. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Για μια ακόμη φορά κατέστησα αφές ότι οι εξαγωγές όπλων είναι ένα άκρο πολύπλοκο ζήτημα. ανθρωπιστικής, ε, ηθικής γεωπολιτικής λοιπά ε, χρειάς. Δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε νωρίτερα στη συζήτηση ο Μίχαλ Γκάλερ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με όλους τους άλλους εξαγωγείς έχει το καλύτερο, το πιο στέρεο σύστημα για την εποπτεία, για τον έλεγχο περιλαμβάνοντα αυτόν τον κατάλογο με κριτήρια. Και κατά πάσα πιθανότητα είναι πρωτοπόρο σε όλο τον κόσμο σε σχέση με αυτό. Και αυτό δεν είναι κάτι που ίσω όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι, αλλά είναι γεγονός. Όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Στο κοινοβούλιο εδώ τουλάχιστον υπάρχουν δύο ομάδες ερωτήσεων κυρίως. Η πρώτη αφορούσε τις εξαγωγές όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα σε χώρες όπως Συρία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Εμένη. Εγώ αναφέρθηκα στα κριτήρια. Το υπαριθμόν 2 κριτήριο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει χρησιμοποιηθεί ως λόγος άρνησης χορήγησης μια σκιάδα εξαγωγών για 72 περιπτώσεις το 2015 και 89 περιπτώσεις το 2016. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Υπάρχει όμως η τάση αυτή που μπορούμε να παρατηρήσουμε, σε ό,τι δεν αφορά. Τις εκκλήσεις για εμπάργκο στην ε, έκδοση άδειας εξαγών για οποιαδήποτε ε, συγκεκριμένη χώρα του κόσμου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απαιτείται ομόφωνη υποστήριξη από όλα τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Τώρα θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ χρήσιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων και να πω ότι ένα από τα βασικά επιτέγματα της κοινή θέση του Βουλή είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά θέματα που από εξαγωγών όπλων. Και η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Το γεγονό ότι οι εθνικέ αποφάσει για τι εξαγωγέ όπλων είναι αντικείμενο αναφορών. Άρα μπορεί κανεί να τα εξετάσει και να τα θέσει από αμφισβήτηση. Ε, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη των αρχών. Αυξάνεται και η λογοδοσία. Έχουμε λοιπόν υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι ο βασικό άξονα. Και αυτά προβλέπει η συνθήκη για τις καλλιέργειες όπλων. Οι αποφάσεις για την χορήγηση αδειών παραμένουν στη δεκτική ευχέρεια των κρατών μελών. Αυτό λέγεται σαφώς. Υπάρχει λοιπόν η εθνική ευθύνη. Η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει τη μεγαλύτερη σύγκληση με ορισμένα κοινά στοιχεία και ανταλλαγή πληροφοριών. Η σύγκληση εξορισμού είναι σίγουρα κάτι που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη. Οι βελτιώσεις που αποφασίστηκαν μετά την αναθεώρηση της κοινή θέση της Ένωσης στηρίζουν την περισσότερη σύγκληση. Σίγουρα ο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο όπω ε, ζητά και η έκθεση μπορεί να δώσει περισσότερα κίνητρα για μεγαλύτερη σύγκληση ολοκληρώνοντα επειδή πρόκειται για κοινά συμφέροντα, κοινά ενδιαφέροντα, θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο το ρόλο του Κοινοβουλίου που διατηρεί ψηλά στην ατζέντα αυτό το θέμα. Το πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε τώρα στην εισηγήτρια, την κυρία Ποντήλ Βαλέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση κατέδειξε πραγματικά πόσο, ε, πόσο διάσταση απόψεων υπάρχει για αυτό το θέμα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βανόρντεν που ανέφερε ότι δεν μιλούμε για τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή τη χρονική ε, συγκυρία. Μιλούμε όμως για την ευρωπαϊκή εμπειρία σε ό,τι αφορά την εξαγωγή όπλων και γι' αυτό στεκόμαστε ε, στην, εξαγωγή όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλούμε για ε, παρεμπόδιση ή απαγόρευση ε, των εξαγωγών, ούτε στερούμε από κάποια χώρα το δικαίωμα να αμυνθεί. Γιατί πολλοί αυτό είπαν από ό,τι φαίνεται. Σας καλώ λοιπόν πραγματικά να διαβάσετε και πάλι την έκθεση πριν ψηφίσετε αύριο. Ανέφερα ότι υπάρχει αυτή η κοινή θέση που είναι ένα καλό νομοθετικό κείμενο και ε, πραγματικά το πιστεύω αν αξιοποιηθεί σωστά. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλές παραβιάσεις αυτών των κριτηριών βάσει της μελέτης ε, που ε, είχε ζητηθεί, όμως τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι έχουν ακόμα πιο ε, στενά και αυστηρά κριτήρια σε σχέση με την κοινή δήλωση. Και αυτό μας οδηγεί στο εξή ερώτημα. Ισχύει κάτι τέτοιο πράγματι. Από τη Γαλλία αναφέρθηκε ότι ε, η Γαλλία έχει το πλέον αυστηρό κριτήριο. Η Ιταλία λέει το ίδιο και η δική μου χώρα το ίδιο λέει. Δεν έχει σημασία όμω ποιο έχει το πλέον αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων. Ε, το θέμα είναι αν ακολουθούμε το κοινό πρότυπο που έχουμε ορίσει από κοινού. Μπορούμε να έχουμε πλέον αυστηρούς βέβαια αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πιο χαλαρούς κανόνες και απλώς να παραπέμπουμε στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε και τη σύμβαση ε, του, του εμπορίου όπλων, όπου ε, τίθεται και ένα ζήτημα της έμφυλης βίας, το οποίο ε, άπτεται των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ένα κριτήριο όμως που δεν συμπεριλαμβάνεται ρητός, εγώ ελπίζω να συμπεριληφθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Όταν